τη διάθεσή τους. Πιστεύω ότι οι ίδιοι πόροι της Ένωσης είναι μια ευκαιρία να αποκτήσουν μια πηγή και να αξιοποιηθεί αυτός ο φόρος ούτως ώστε να δώσουμε αυτή την όθηση που χρειάζεται η ανάπτυξη στην Ευρώπη. Είναι μια στιγμή δημιουργίας και πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κάνω μια σύντομη ανακοίνωση. Υποκαλωσορίζουμε μέλη του Κοινοβουλίου του Μεξικού στην αίθουσα κάθονται πάνω στα έδρανα των επισκεπτών. Τους ευχόμαστε ευχάριστη διαμονή στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο. Thank you very Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συνεχίζουμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Κάλφιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω ότι θα υποστηρίξουμε ευρέως τη σημερινή ψηφοφορία. Πολλοί ανησυχούν από ό,τι βλέπω για τις επιπτώσεις του φόρου για τους φορολογούμενους και συμφωνώ. Όλοι έχουμε ανησυχίες γι' αυτό. Αλλά σας καλώ να δείτε τι πληρώνουν για την εξυγίανση του οικονομικού, του χρηματοπιστωτικού συστήματος οι πολίτες σε ό,τι αφορά και τις παρεμβάσεις των διαφόρων μηχανισμών εκατομμύρια και δισεκατομμύρια χρησιμοποιούνται για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αν ο φόρος καθιερωθεί, το βάρος για τους φορολογούμενους θα μειωθεί. Όχι πλήρως, αλλά μερικώς. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αν ένα τμήμα διοχετευθεί προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό δεν θα είναι ένα συμπληρωματικό φόρος. Σημαίνει ότι οι εθνικές εισφορές θα μειωθούν, που τελικά σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι τα έσοδα αυτού του φόρου θα καταλήγουν στον εθνικό προϋπολογισμό και αυτό είναι βεβαίως προ το συμφέρον των φορολογούμενων. Η κυρία Γκάλ Πέλτς, επόμενη μιλήτρια θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που περιλαμβάνει η έκθεση η οποία λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι οι συναλλαγές κατά το παρελθόν δεν φορολογήθηκαν επαρκώς και εκτός αυτού η έκθεση είναι ένα κείμενο το οποίο ε, προσφέρει πραγματικά μια λύση για την ευρωπαϊκή κρίση. Εδώ γίνεται το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση της Κρήτης και η έκθεση περιλαμβάνει και πρακτικά αποτελέσματα. Δυστυχώς ο φόρος αυτός δεν μπορεί να επιβληθεί παγκοσμίως ίσως ούτε καν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όμως μπορούν να υπάρξουν σημαντικοί πόροι για την ευρωπαϊκή οικονομία. Η ενισχυμένη συνεργασία είναι ένα καλό εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει στο να ρυθμίζονται ε, ικανοποιητικά οι συναλλαγές και με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος οι συναλλαγές να αποκοπούν πλήρως από την πραγματική οικονομία. Ο τομέας χρηματοψηφικών συναλλαγών είναι εκείνο που προκάλεσε την κρίση διότι είχε κατά νου μόνο τους δικούς του στόχους και δεν συνέβαλε στο να βγει από την κρίση ενισχυμένος. Η έκθεση λοιπόν αυτή εξετάζει ε, τις αντιφάσεις, το πώς είναι δυνατόν να αρθούν οι αντιφάσεις. Η έκθεση συμβάλλει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και επίσης και στο να κλείσουν τα νομικά παραθυράκια ε, και να ε, αποφεύγεται και η φόρα αποφυγή. Ο κύριος Λάχτφριντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι με τον φόρο επί των χρηματοψηφιωτικών συναλλαγών έχουμε στα χέρια μας ένα εργαλείο που επιτρέπει στο μέλλον να κατανέμεται ε, δίκαια το βάρος της κρίσης. Έχουμε ένα εργαλείο που επιτρέπει ακόμα και αυτοί που μέχρι τώρα αρνήθηκαν να καταβάλουν φόρους, δηλαδή οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρήσεων, οι τράπεζες, αυτοί θα πρέπει πλέον να πληρώνουν φόρους. Και έχουμε ένα εργαλείο που προκαλεί ανάπτυξη. Ανάπτυξη εκεί που είναι απαραίτητο. Στην πραγματική οικονομία και όχι στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Νομίζω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο ε, με την ψηφορία τη σημερινή ε, θα επιτύχει τους στόχους του. Βέβαια δεν είμαι ικανοποιημένο με αυτά που γίνονται στο Συμβούλιο. Αυτά που διαδραματίζονται τώρα στο Συμβούλιο είναι σκάνδαλο. Ο κύριος Κάμερον και οι όλο και λιγότεροι φίλοι του κατορθώνουν τελικά την πολιτική τους να τη στρέφουν προς δισεκατομμυριούχους και αυτοί να την επιβάλλουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, στον κύριο Κάμερον και στους φίλους του στο Συμβούλιο ας τους δώσουμε σήμερα την απάντησή μας, ας ψηφίσουμε υπέρ του χρηματοψηφικού φόρου εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Κάρας. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ισηγήτρια, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σημερινή έκθεση για άλλη μια φορά ε, τεκμηριώνει το ότι διαδραματίζει πρωταρχικό και ε, σημαντικό ρόλο, το ρόλο του σκαπανέα στο φόρο επί των χρηματοεπιστωτικών συναλλαγών. Το Κοινοβούλιο με αυτή την έκθεση αποδεικνύει και το ρόλο σκαπανέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και οι προλαλήσαντες και εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο μπλοκάρει μια πανευρωπαϊκή εισαγωγή του φόρου. Το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή μπλοκάρει την ε, εισαγωγή ε, του φόρου αυτού στο σύνολο της Ευρωζώνης. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο καθιστά μη ρεαλιστική την εφαρμογή αυτού του φόρου. Γιατί αν μόνο εννέα κράτη είναι υπέρ αυτού του φόρου, καταλαβαίνετε ότι ο φόρος αυτός μπορεί να αποδειχθεί και μειονέκτημα. Εμείς θέλουμε να σπάσουμε το μπλοκάρισμα, τον αποκλεισμό για μας ο φόρος αυτός είναι μέτρο πολιτικής τάξης και επειδή είναι μέτρο πολιτικής τάξης για το λόγο αυτό εγώ κατέθεσα τροπολογία με βάση την οποία οι συναλλαγές πέρα από τις χρηματιστηριακές πρέπει να φορολογούνται περισσότερο από τις ενδοχρηματιστηριακές. Εμείς ε, το φόρο αυτό θέλουμε να τον χρησιμοποιήσουμε, να υπάρχουν περισσότερα έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Παρακαλώ να υπερψηφίσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σήμερα πριν από την ψηφοφορία της έκτησης ε, Ποδηματά ήρθε η στιγμή να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, είναι απαραίτητος αυτός ο φόρος. Εκ των όνου Είναι η μόνη στρατηγική εξόδου από την κρίση που μπορεί να υπάρξει. Εγώ ε, το λέω ως Αυστριακή η οποία είναι υπέρ αυτού του φόρου. Η κερδοσκοπία είναι επικίνδυνη, είναι εκείνη η οποία προκάλεσε τα δεινά και την κοινωνική κρίση. Αν θέλετε ήταν και το αίτιο της κρίσης. Οι τράπεζες πρέπει να σώζονται. Αυτό συμβαίνει καθημερινά. Η Ευρώπη βυθίστηκε σε κρίση. Ε, γι' αυτό λοιπόν τώρα και όχι στο απότερο μέλλον καλούμεθα να εγκρίνουμε το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, πληρώνουμε φόρους για τα πάντα, για την εργασία, την ενέργεια. Είναι παρά παράλογο ο φόρος χρηματοψηφιακών συναλλαγών να μην έχει ήδη εισαχθεί. Προσβλέπω λοιπόν από αυτό το φόρο μεγαλύτερη σταθερότητα των αγορών, περιορισμό της βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπίας και κυρίως μεγαλύτερο εστιασμό στην πραγματική οικονομία ή αν θέλετε χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Δεχάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, ακούσαμε ήδη πολλές φορές στη συζήτηση, η θέσπιση ενός τέτοιου φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι εύλογη εφόσον έχει μία ευρωπαϊκή διάσταση, δηλαδή εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν γίνεται τουλάχιστον να έχει παγκόσμια διάσταση που θα ήταν το καλύτερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει έναν ευρωπαϊκό φόρο. Οπότε το επόμενο λογικό βήμα θα ήταν να έχουμε και ευρωπαϊκού ίδιου πόρου, με ευρωπαϊκά έσοδα, ώστε να έχουμε μια στέρεη βάση στον προπολογισμό μα, όπω ισχύει για του εθνικού προπολογισμού. Επιπλέον, έτσι θα μπορούσαμε να τονώσουμε την ανάκαμψη ε, και την ανάπτυξη, γιατί με έναν φόρο τέτοιο και κοινοτικά έσοδα θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε όλα τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στην έκθεση Λαμασούρ και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε δηλαδή να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που θα είναι εργαλείο για την ανάκαμψη και την τόνωση της ανάπτυξης. Έτσι θα μετριάσουμε κάπως το βάρος και των εθνικών προϋπολογισμών. Έχουμε λοιπόν ένα σημαντικό εργαλείο που επιτελεί ταυτόχρονα ένα διπλό στόχο και τα οικονομικά και τονώνει την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμασούρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συζήτηση που διεξάγεται, γιατί κάθε εβδομάδα ακούμε αριστερά και δεξιά κάποιους πολιτικούς ευθύνοντες να υποβάλλουν τις προτάσεις, λες και ήταν ε, επαναστατικές προτάσεις και δική τους ε, ιδέα και φαϊνή. Ενώ πριν από πέντε χρόνια είχαμε μια τέτοια θετική στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πριν από ένα χρόνο είχαμε συγκεκριμένο περιεκτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σεμέτα. Και μάλιστα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, εργάζεται εδώ και έξι μήνε για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι ε, ο φόρος αυτός είναι έμεσος φόρος όπως ο ΦΠΑ. Μην ε, έχουμε αυταπάτες για τη φύση του και επιβάλλεται στα, στους χρηματοπιστωτικούς φορείς, αλλά με τέτοια ευρεία φορολογική βάση και με τέτοιο χαμηλό φορολογικό συντελεστή που θα είναι ανεπαίσθητη η επιρροή του. Ε, ούτε θα έχει ως αποτέλεσμα την μετεγκατάσταση χρηματοπιστωτικών φορέων. Άλλωστε είναι και διπλός ο στόχος αυτού του, στόχου, του φόρου, χρηματοδότηση των ε, κοινοτικών στόχων και ε, ελάφρυνση των εθνικών προϋπολογισμών. Βέβαια η ομοφωνία θα είναι δύσκολη στο Συμβούλιο, αλλά αν καταλήξουμε στη συμφωνία ώστε να έχουμε παρόμοιο φόρο σε σημαντικό αριθμό των χωρών μελών, είναι σημαντικό είναι φυσιολογικό τα έσοδα να πηγαίνουν στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Έτσι θα μειώνονται οι εθνικές συνεισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό και τα κράτη-μέλη θα ανακτήσουν περιθώριο λιγμών για να μειώσουν και το δημόσιο χρέος τους και το έλλειμμά τους. Και όσοι δεν τον προσυπογράψουν, δικό τους ε, ε, χάσιμο και σφάλμα. Ο κύριος, ο κύριος Κάσα, επόμενος ομιλητής. Η συμπεριφορά αυτή του χρηματοπιστωτικού τομέα οδήγησε στην κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Συνεπώς πρέπει να κληθεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας να πληρώσει το τίμημα. Δεν πιστεύω ότι ο φόρος αυτός είναι όμως ο σωστός τρόπος να λυθεί το πρόβλημα, διότι το κόστος του φόρου θα μετακυλιστεί στους καταναλωτές και είναι επικίνδυνο για την Ευρώπη να πιστεύουμε ότι καθιερώνοντας ψηλά πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι θα κάνουν το ίδιο και άλλες δικαιοδοσίες δεδομένης της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε πρέπει να εξασφαλίσουμε έναν υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα που και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ε, όταν σκεφτόμαστε να καθιερέσουμε ένα φόρο ή μια πολιτική που μπορούν να μην οδηγήσουν στον σκόπο που επιδιώκουμε. Αρχικά είχαμε μιλήσει για σημαντική μείωση του ΑΕΠ. Μετά από κάποιες κριτικές προσάρμοσε την αξιολόγησή της η Κομισιό για να αποδείξει το αντίθετο. Λόγω αυτής της κατάστασης δεν υποστηρίζω την καθιέρωση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλώ τους συναδέλφους να με υποστηρίξουν ψηφίζοντας κατά της πρότασης της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κυρίες και κύριοι θα κάνουμε μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα. Λόγο διότι η Υπουργό Φεστάρ πρέπει να, να χωρίσει. Πριν από το Catch the Eye, λοιπόν, θα της δώσω το λόγο εξ ονόματος του Συμβουλίου. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση που έδειξε σαφώς ότι η δουλειά που έχει ήδη γίνει στα πλαίσια της παρουσίασης της Επιτροπής για τον φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ήταν σημαντική. Οι τρισχιώδεις εισηγητές έκαναν πολύ καλή δουλειά και έγινε και πολύ καλή δουλειά και στις διάφορες επιτροπές του Κοινοβουλίου. Μιλάμε για ένα φάκελο που επανέρχεται και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τον συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου. Το καθαριστικό παράγοντας σημερινή συζήτησης είναι η ομοφωνία που διαπιστώθηκε για την ανάγκη ε, να έχουμε ένα χρηματοπιστωτικό τομέα ο οποίος λειτουργεί αποτελεσματικά, κάτι σημαντικό για την ανάπτυξη και χρειαζόμαστε έναν τέτοιο τομέα ο οποίο θα στηρίζει τα υγεία προϊόντα ενώ θα αναλαμβάνει, χωρίς να αναλαμβάνει κινδύνους ώστε να μην μπορούν να αποκτήσουν τις πιστώσεις που χρειάζονται οι καταναλωτές. Ευχαριστώ όλους για τη δουλειά που έγιναν από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το πρώτο αυτό αποτέλεσμα που οφείλεται στις ε, εργασίες των προηγούμενων προεδριών ήταν μια ανάλυση για τα παράγωγα προϊόντα. Και αυτή είναι μια και αυτό ήταν ένα σημαντικό βήμα. Ακολούθησε η απόφαση του Συμβουλίου των τελευταίων ημερών, η οποία θα μας επιτρέψει να έχουν μεγαλύτερη ανεξαρτησία των οίκων αξιολόγησης και αυτό θα επιτρέψει επίσης μία ε, τελική απόφαση για το πώς θα γίνεται η αξιολόγηση των πιστώσεων. Ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να προβλέψει μια συζήτηση εδώ για τα project bonds και δεν είναι όμως αυτό το πιο σημαντικό. Πρέπει επίσης να ξεκινήσει η τριμερή συνομιλία για τα κεφαλουχικά έργα. Η Επιτροπή έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις για τη ρευστότητα, την ποιότητα του κεφαλαίου, ε, αυτά που ε, πραγματοποιούνται και ο τρόπος με τον οποίο εξασφαλίζουμε ότι ως χρηματοπιστωτική επιχείρηση να συμπεριφερθούμε προτού να ε, καταβάλουμε μερίσματα. Η σημερινή συζήτηση μας επέτρεψε να μιλήσουμε για ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών. Αλλά απαιτείται ομοφωνία σε επίπεδο Συμβουλίου. Διότι έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα στο Συμβούλιο που είναι η καλύτερη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα και αυτό είναι σημαντικό. Η συζήτηση για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών συμπληρώνει μια ημερήσια διάταξη σημαντική για το θέμα της ρύθμισης. Ε, τέθηκαν σειρά ερωτημάτων σήμερα από τα μέλη του Κοινοβουλίου που υποστηρίζουν τον φόρο ή εκείνων που είναι κατά αυτού του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Πώς θα λειτουργήσει, πώς θα εφαρμοστεί γνωστή, θα ε, πληρώσει το λογαριασμό, θα, θα υπάρξουν απαλλαγέ για ορισμένους, υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε κερδοσκοπική και μη κερδοσκοπική συναλλαγή, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας ενισχυμένη συνεργασία. αν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης ομοφωνίας στο Συμβούλιο. Πάρα πολλά μέλη τόνισαν ότι θα, υπάρξει, θα είναι δύσκολο να προκύψει ομοφωνία στο Συμβούλιο και πιστεύουν ότι θα ήταν προβληματικό να, υπάρξει, να έχουμε για την εσωτερική αγορά ενισχυμένη συνεργασία. Τέλος, και αυτό παραμένει σημαντικό, αυτή η συζήτηση αφορούσε τη διάθεση των πόρων. Επίσης, στο Συμβούλιο θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας πάνω σε αυτό το θέμα λάβαμε γνώση και τη σημερινή συζήτηση και των προτάσεων του Κοινοβουλίου που επιθυμεί η δουλειά αυτή, οι εργασίε να συνεχιστούν. Ακολουθούμε δύο κατευθύνσει, όπω σα είπα. Εξετάζουμε την πρόταση τη Επιτροπή αφενό και η σημερινή συζήτηση συμβάλλει σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα συνεχίζουμε και τι εργασίε μα για εναλλακτικέ προτάσει που θα μπορούσαμε να υποβάλουμε για, αντί αυτού του φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Υπάρχουν στι διάφορε χώρε διαφορετικοί φόροι, το τέλο χαρτοσύμου που αναφέρθηκε πολλέ, ο φόρο επί των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που επίσης υπάρχει. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλες για αυτή τη συζήτηση που ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ζωντανή και τη συμμετοχή και τη συνεισφορά σας στις εργασίες του Συμβουλίου επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε το έργο μας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο και ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Σας εύχομαι και καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Πέραμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε τριπλάσιο αριθμό αγορητών, τουλάχιστον ε, επίδοξων αγορητών. Δεν μπορώ να ικανοποιήσω δυστυχώς όλους τους συναδέρφους. Θα περιορίσω τον αριθμό των ε, μιλητών. Ο πρώτος είναι ο κύριος Κέλλη στο Catch the Eye. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε χρέο. ψάχνουμε να κερδίσουμε τα κενά με τους φόρους και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο φαινόμενο φοροαποφυγής. Βέβαια, εδώ ο κόσμος καίγεται ε, και φαίνεται ότι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς κερδίζουν ενώ οι πολιτικοί χάνουν ε, το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Στο G20 ζητήσαμε ε, παγκόσμια εφαρμογή του φόρου αυτού, ώστε καμία χώρα να μην κερδίσει βάρος των άλλων. Μία ίσον σημασία βέβαια πρόταση, μια δεύτερη σε αξία πρόταση είναι τουλάχιστον να εφαρμόσουμε στις 27 χώρες μέλη. Θα μπορούσαμε μεταβατικά σε 2-3 χρόνια να το εφαρμόσουμε και να δούμε τι προβλέψεις και τι συνέπειες έχουμε για μετακαταστάσεις. Εγώ πολύ αφιβάλλω. Γιατί επαναλαμβάνω τόσο ε, μικρή η φορολογική συντελεστές 0,1 και 0,01 που δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τέτοια μετακατάσταση. Η κυρία Ταμπάιτζη. Ο κύριος Ταμπάιτζη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δυστυχώ υπάρχει κάποιο... Ναι, υπήρχε πρόβλημα το οποίο λύθηκε. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να μετακυλήσει το κόστος της κρίσης στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Ε, πρόκειται για ε, κερδοσκόπες ε, συναλλαγές που πρέπει να φορολογηθούν και με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι θα υπάρχει δικαιότερη αντιμετώπιση της κρίσης. Η Ουγγρική κυβέρνηση όμως ε, μοιάζει να θέλει να φορολογήσει ή να επιβαρύνει τους ε, καταναλωτές. Η δική μας η κυβέρνηση ε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό το φόρο για τον οποίο συζητάμε σήμερα. Οι πολίτες θα επιβαρυνθούν οι τραπεζικές συναλλαγές, τα εμβάσματα, όλα αυτά ε, θα επιβαρυνθούν. Θέλω να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να φορολογήσουμε τους ε, ολιγάρχες και τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η κυρία Μιράντα. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ. Κυρία Ποδηματά. Είναι πολύ χρήσιμη, αξιέπαινη προσπάθειά σας, πολύ αξιόλογη. Ε, χρειαζόμαστε ε, πραγματικά τόλμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε την κερδοσκοπία στο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι ένα πολιτικό μήνυμα που περιμένουν όλοι οι πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε μια πορεία για να αποσοβήσουμε την εγκληματική μερικές φορές κερδοσκοπία των χρηματοπιστωτικών φορέων. Θέλουμε αυτός ο φόρος ε, να περιορίσει αισθητά την κερδοσκοπία. Είναι πολύ χρήσιμος επίση για να ε, τονώσουμε την επενδυτική δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκής Ένωση να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση, να αποκαταστήσουμε τη διαφάνεια, να διενεργήσουμε καλύτερους ελέγχου και να επιβάλλουμε κυρώσει κατά κάποιο τρόπο στις κερδοσκοπικές δραστηριότητε. Είναι πολύ δυστυχώ αυτοί που πλήττονται από την τραπεζική χρεοσκοπία μέσω τη ε, συμμετοχή. ή ε, προτιμησιακών ομολόγων, ανθρώπων που επενδύουν ε, τους ε, μισθούς και τις αποταμιεύσεις και δεν μπορούν δυστυχώς να έχουν καμία απόδοση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγητρία. Κυρία Αντζελίλη, σήμερα το Κοινοβούλιο μπορεί να δώσει ένα χειρό μήνυμα στο Συμβούλιο έτσι ώστε να εισάγει το χρηματοψηφιακό φόρο. Κυρίω ένα μήνυμα σαφέ προ του πολίτε και τι επιχειρήσει που μα ρωτούν μα τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση. Εξ ονόματο λοιπόν της Αθήνα ο φόρος επί των χρηματοψηφιακών συναλλαγών θα αποδώσει περίπου 60 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να διοχετευτούν στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην ε, συγκράτηση της φορολογικής πίεσης επί των πολιτών. Όμως θα είναι και ένα μήνυμα ισότητα δικαιοσύνης, διότι ο τομέας, ο χρηματοψηφιακός, το ζητάνε οι πολίτες, πρέπει και αυτός να συμβάλλει έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το κόστος της οικονομικής κρίσης. Και ο τομέας αυτός πρέπει να αναλάβει τις του. Ευχαριστούμε την κυρία Ποτηματά για τη στράτευσή της για το θέμα αυτό. Επόμενη η κυρία Φλασίκοβα Μπένοβα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα το Κοινοβούλιο με την ψηφοφορία και το Κοινοβούλιο με την ψήφο του θα στείλει ηχηρό μήνυμα όχι μόνο προς το Συμβούλιο αλλά και προς τους πολίτες γιατί μέχρι τώρα οι πολίτες είναι εκείνοι που καλούνται να καλύψουν ε, τα χρέη του χρηματοψηφιακού τομέα. Ο φόρος αυτός μπορεί λοιπόν να καταστεί πολύ σημαντικός για την αντιμετώπιση της κρίσης, όχι μόνο σε μεμονωμένα κράτη-μέλη Ο φόρος αυτός μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σύνολο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν σημαντικό να σκεφτούμε, να δούμε πώς μπορεί να επιμεριστεί ο φόρος αυτός και πώς μπορούν να περιοριστούν οι δαπάνες για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Μέχρι 70 δις ευρώ μπορούμε να ε, κερδίσουμε και να ενισχύσουμε την εσωτερική αγορά. Ε, με το φόρο αυτό θα αμπληνθούν οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και θα αποθαρρυνθούν οι κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Μεσάρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η οικονομική κρίση εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην πραγματική οικονομία και αυτό έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην απασχόληση. Οι διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έκαναν πάρα πολύ σοβαρές και βαριές περικοπές και ο χρηματοπιστωτικός ε, τομέας έλαβε πάρα πολλές κρατικές ενισχύσεις, χωρίς από την πλευρά του να συνεισφέρει στην ε, υπέρβαση της οικονομικής κρίσης ή να προλιάνει τουλάχιστον το έδαφος για να βγούμε κάποια στιγμή. Η οικονομική κρίση και ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που μας απασχολούν. Μπορούν έτσι να μετριαστούν οι διάφορες κερδοσκοπικές δραστηριότητες και τα έσοδα να φτάσουν ε, σε 57 ε, δισεκατομμύρια ευρώ για να ε, επιμεριστεί το κόστος και το βάρος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εισαχθεί αυτός ο φόρος είναι πολύ μεγάλο κέντρο χρηματοπιστωτικό η Ευρώπη και αυτό είναι πρώτο βήμα. Κύριε Λιμπεράτσικη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άννη Ποδηματά, να τη συγχαρώ θερμότατα για την πολύ αξιόλογη έκθεσή της. Και με πολύ μεγάλη ικανοποίηση δεχόμαστε και την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φαίνεται ότι αρχίζει νέα πνοή και στο Συμβούλιο και θα ήθελα να παροτρύνω την Δανική Προεδρία να προσπαθήσει να ευθυγραμμίσει το Συμβούλιο με την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχουν βέβαια διαστασίες απόψε σε πολλά κόμματα και στο δικό μας. Ακούσαμε μερικές ομιλίες που ήταν πολύ περιπτωσιολογικές γιατί αναφερόταν τα παραδείγματα της Ολλανδίας, της Σουηδίας. Παρ' αυτά Πιστεύω ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε ε, και ε, ενώ θέλουμε να εξοικονομήσουμε εκατομμύρια, δεν έχουμε την ευκαιρία να εισπράξουμε δισεκατομμύρια. Και με τέτοια τεράστια κονδύλια μπορούμε να ενισχύσουμε την ανάπτυξη, να δημιουργήσουμε νέε θέσει απασχόληση, να αφιερώσουμε αυτά τα θέματα για νέε αναπτυξιακέ ε, δυνατότητε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζούμπερ. Ευχαριστώ. Από το τέλος δεκαετίας του 1990 ζητούμε ένα φόρο επί το χρηματοπιστωτικό συναλλαγών στο χρηματιστήριο. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για να, για πατάξουμε την κερδοσκοπία. Είναι ανεπαρκές όμως αυτό το εργαλείο. Χρειαζόμασταν πιο θαραλέα και τολμηρά μέτρα. Για παράδειγμα, τέλο στου φορολογικού παραδείσου και τα πιο κερδοσκοπικά χρηματοπιστωτικά παράγωγα. Αυτό θα ήταν η κατάλληλη λύση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και ο φόρο αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Η πρόταση αυτή, βέβαια, αφορά, δίνει πιο ευνοϊκή μεταχείριση στα παράγωγα και τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δίνοντα ένα πολύ χαμηλό συντελεστή, 0,01%. Πολύ πιο προνομιακό. Πιστεύω πάντως ότι τα έσοδα αυτού του φόρου θα πρέπει να αφιερωθούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και να μην ελαφρύνουν τις εθνικές συνεισφορές στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Βέβαια, ούτως ή άλλως έχουμε χαμηλή συνεισφορά και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να ενισχύσουμε τα ταμεία σύγκλησης και κοινωνικής συνοχής. Ευχαριστώ και για τα τελικά σχόλια. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Σεμέτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, Υπουργέ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την μεγάλη υποστήριξη ε, για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό μήνυμα προς τα κράτη-μέλη. Συνεχίζονται οι συζητήσεις στο Συμβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δανική Προεδρία που διατηρεί ε, αυτή ε, τη συγκυρία και την ορμή στη διαδικασία και των τεχνικών συζητήσεων. Το Μάρτιο στο άτυπο Συμβούλιο Κοφίν συμφώνησαν οι Υπουργοί να συνεχίσουν τα εργαστήρια ε, που επεξεργάζονται την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή τη βάση, ε, βράχει πρόθεσμα θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτάσει που ενδέχεται περισσότερο να ευδοκιμήσουν. Καλωσορίζω την πρόταση τη Δανική Προεδρία που προτίθεται στι 22 Ιουνίου στο ΕΚΟΦΗ να κάνει μια προσανατολιστική συζήτηση. Στο μεταξύ θα εξακολουθήσω να υποστηρίζω ε, ένα ευρύ φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε για ε, να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική και η ανάπτυξη και να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν ισόρους παιχνιδιού. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ αυτού του φόρου και είναι σωστά όλα. Επίσης, ακούσαμε και κάποιες ανησυχίες για συγκεκριμένα επιμέρους σημεία. Χρειάζεται περαιτέρω τεχνική επεξεργασία από εμπειρογνώμονες των κρατών μελών που θα επιφέρει και σαφήνεια και λύσεις. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή. Θα ήθελα γενικά να τονίσω το εξή. Ο φόρος επί το χρηματοπιστωτικό συναλλαγό θα βοηθήσει να κατασταθεί η ε, σχέση μεταξύ του χρηματοπιστωτικού ε, τομέα και του απλού πολίτη. Να αποκατασταθεί λέγω αυτή η σχέση που έχει ε, πληγεί τα μάλα τα τελευταία έτη. Έτσι θα στραφεί προς την πραγματική οικονομία περισσότερο ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Θα βοηθήσει αυτός ο φόρος για την ατζέντα της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Ποδηματά. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, αγαπητοί συνάδελφοι, για να είμαστε συνεπείς στις θέσεις μας, υπενθυμίζω ότι στην Ευρώπη ήδη εννέα χώρες έχουν ε, μια, ε, έναν ανθυρό τέτοιο κλάδο με χρηματοπιστωτικά ε, κέντρα που υπόκεινται στο φόρο και είναι ανθυρά. Άρα λοιπόν η επιβολή του FTT δεν οδηγεί σε μετεγκατάσταση των χρηματοπιστωτικών ε, ιδρυμάτων. Επίσης Κάποιοι συνάδελφοι εξέφρασαν φόβους για τα αρνητικέ επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά από το φόρο. Η αλήθεια είναι ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις τώρα υποφέρουν λόγω της χρηματοοικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από το χρηματοπιστωτικό τομέα λόγω των υψηλών επιπέδων ΦΠΑ και των υψηλών ε, φόρων στην εργασία. Για τις ε, εξαιρέσεις συμφωνώ με τον Επίτροπο Σέμετα ότι οι εξαιρέσεις δημιουργούν παραθυράκια και στρεβλώσεις. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην Επιτροπή ΕΚΟΝ, στα πλαίσια της Επιτροπής Οικονομικών Νομισματικών Υποθέσεων, καταλήξαμε σε μια συμβιβαστική λύση μέχρι την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας, με πνεύμα συμβιβαστικό που λυπάμαι που δεν επιδεικνύεται επαρκώς, παρά το γεγονός ότι η FTT θα επηρεάσει ελάχιστα τα συντηρητικά κεφάλαια και αντίθετα μπορεί να διασφαλίσει καλύτερα τι συντάξει των Ευρωπαίων, δίνοντα κίνητρα για να ακολουθούν σόφρονες επενδυτικές στρατηγικές. Αν όμως ε, ζητήσουμε περισσότερες εξαιρεσει σε επενδυτικά προϊόντα, που μπορεί να ε, έχουν ρίσκο στην επενδυτική τους πολιτική, αυτό νομίζω ότι δεν θα συνάδει με τον στόχο που επιδιώκουμε. Συμπεραίνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας καλέσω να εγκρίνετε με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση ε, για τον ε, φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών αποστέλλοντας ένα ισχυρό μήνυμα προς το Συμβούλιο ιδιαίτερα σήμερα στο φως της άτυπης Συνόδου Κορυφής ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ανάπτυξη και να επιβεβαιώσουμε ότι το Κοινοβούλιο αυτό ήταν και εξακολουθεί να είναι συνεπές με τις μεγάλες πολιτικές και προσεγγίσεις που υποστήριξε από την αρχή της εκδήλωσης της κρίσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η ε, συζήτηση και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο θέμα μας ε, είναι συζήτηση